Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία ε, Ένταξης ε, του Κωσφοπεδίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον Υπουργό κύριο Κιόντερς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ε, χαιρετήσω την πρόσφατη συμφωνία της σχέση σας, τη σταθεροποιημένη σχέση με το Παιδί. Τώρα πλέον να πω και το Συμβούλιο να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να τη θέσει σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η διαδικασία σταθεροποίησης ε, και ε, διασύνδεση ένωση με το Κωσοπέδιο, κατά την άποψή μου, είναι ένα σημαντικό μήνυμα, μήνυμα υποστήριξη και πολύ καθοριστικό, μεγάλη σημασία για το Κωσοπέδιο. Ξερτάται βέβαια το πώ θα εφαρμοστεί η συμφωνία. Οι άνθρωποι στο Κοσμοπέδιο πρέπει να αισθαντούν τα συγκεκριμένα ωφέλη από τη συμφωνία εάν υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Εναπόκειται λοιπόν στο Κοσμοπέδιο να εστιάσει την προσοχή του στην εφαρμογή της ε, συμφωνίας στο κράτος δικαίου, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης πάνω απ' όλα. Το κοσφοπέδιο πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, μεγάλο πρόβλημα, και ε, να προχωρήσει και άλλες υποθέσεις που εκκρεμούν στη δικαστική οδό. Κατά την άποψή μας ε, υπάρχουν θέματα στο κοσοπέδιο που ε, πρέπει να επιληθούν ταχύτατα. Καταδικάζουμε τη βία από όλε τι πλευρέ ε, γιατί η λύση είναι ο πολιτικό διάλογο. Κατόπιν τούτου πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για τι μεταρρυθμίσει στο κοσοπέδιο. Ουσιαστική πολιτική βούληση απαιτείται από όλου του εμπλεκόμενου για να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη εσωτερική κατάσταση και για να προχωρήσει το κοσοπέδιο. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασικό συστατικό για να σταθεροποιηθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Η σταθεροποίηση και η σύνδεση συμβαδίζουν χέρι-χέρι και η σταθεροποίηση σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει και η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία. Αυτό το συζητήσαμε και προηγουμένως. Αν δεν υπάρξει σταθεροποίηση, ορατή, ε, θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενθαρρυντικές ήταν οι εξελίξεις πέρυσι ε, στον διάλογο και διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν ήταν εύκολο πολιτικά. Εξακολουθεί και παραμένει ένα ευαίσθητο πολιτικά θέμα. Ένα θέμα που διχάζει Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για το Κοσμοπέδιο το, σημαντικότερο δυνατό, το συντομότερο δυνατόν να εφαρμόσει τη συμφωνία παρά τις εσωτερικές δυσκολίες. Και γι' αυτό η συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στους Μούσταφας και Μπούτσιτς εγώ ενθαρρύντηκα γιατί εκεί επιβεβαιώθηκε η σημασία του διαλόγου και για τις δύο χώρες. Το Συμβούλιο παρακολουθεί τις εξελίξεις εκ του Σύνεγγης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Κοσμοπέδιο. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις κοινωνικέ μετα μεταρρυθμίσει στο Κωσυφοπαίδιο μέσα από οικονομική και τεχνική αρρωγή. Η οικονομική ανάπτυξη είναι εκείνη ε, που υπολείπεται η βελτίωση οικονομίας είναι βασικό πρόβλημα στο Κωσυφοπαίδιο. Και να πω και κάτι άλλο για τη διαδικασία Απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων. Πολύ σημαντικό για το κοσυφοπαίδιο. Η Κομισιόν ε, είπε πρόσφατα ότι το κοσυφοπαίδιο προχωράει σταθερά σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Αναφέρει βέβαια εννέα εκκρεμούσες προϋποθέσεις ε, για τέσσερις σημαντικούς τομείς. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό για το κοσμοπέδιο να ε, επιληφθεί αυτών των θεμάτων από τη στιγμή που θα, έχουν, θα τα κριτήρια το, θέμα θα, το Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα. Και τέλος να ε, υπογραμμίσω πόσο σημαντική είναι η Ulex, η οποία στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις και το κράτος δικαίου στο Κωσυφοπαίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να πάρει το λόγο ο κύριο Χάν, παρακαλώ, πλευρά της Επιτροπής. Κύριε Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι, πριν από δύο εβδομάδε ε, σα μίλησα εδώ για να σα ευχαριστήσω για τη στήριξή σα στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη των σχέσεων μα με το κοσμοπέδιο και τη στήριξή σα για την ε, συμφωνία σταθεροποίηση και σύνδεση που διαπραγματοποιήκαμε με το κοσμοπέδιο. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΑΦΕΤ και ιδιαίτερα την εισηγήτρια Ουλή και Λίνατσεκ για τη στήριξή τη. Το σώμα σα στήριξε με δύο πλειοψηφίε για τη στήριξη αυτή τη συμφωνία στι 24 Ιανουαρίου. Και αυτό έγινε δεκτό με ικανοποίηση και στι Βρυξέλλε και στην Πρίστινα. Και αυτό θα επιτρέψει και εμά να εγκρίνουμε αργότερα μέσα στο μήνα τη συμφωνία αυτή και αυτό καταδεικνύει την στήριξη που έχει το Κωσοπέδιο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αρχίσουμε την εφαρμογή τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία μόνο θα εμβαθύνει τι πολιτικέ μα θέσει, θα διασφαλίσει μια πιο προβλέψιμη διαδικασία ανάπτυξη των σχέσεων για να έχουμε ε, απασχόληση και να ελπίζουμε πολιτική πολιτική ηγεσίε που καταφέρει να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία, την έγκριση δηλαδή αυτή τη συμφωνία σταθεροποίηση και σύνδεση για να συζητήσουμε γύρω από ένα τραπέζι τι διαφορέ του για να φύγουμε από το πολιτικό αδιέξοδο. Αυτή η πολιτική παράλυση στο Κοσμοπέδιο, στην Πρίστινα, έχει κρατήσει πάρα πολύ και έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Πρέπει επιτέλου η αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τη βία και την παρακόλληση και να αρχίσει να εργάζεται σοβαρά. Η έκθεσή μα ε, για το Κοσμοπέδιο του 2015 ότι το Κοσμοπέδιο πρέπει να επιβάλλει σε τομεί κλειδιά. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανεργία που είναι πολύ ψηλή και η οικονομική ανάπτυξη ανεπαρκής. Πρέπει να εστιαστεί περισσότερη προσπάθεια στην επίτευξη αποτελεσμάτων, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διαφορά. Και το αυτό ισχύει για την εξαρτησία και τη δυνατότητα δράση ε, του δικαστικού τομέα. Οι δράσει σε αυτού του τομεί θα χορηγήσουν στου πολίτε του Κοσμοπεδίου μια ευρωτική καλύτερου όπως αναφέρει και η συμφωνία, αποδίδουμε τεράστια σημασία στην εξομάλυνση των σχέσεων του Κόσμου Παιδίου με τη Σερβία. Το σκοπέδιο πρέπει να εφαρμόσει τι συμφωνίε τι οποίε έχει καταλήξει και να συνεχίσει να εργάζεται προ περαιτέρω συμφωνίε. Το Κοσμοπέδιο πρέπει επίση να διασφαλίσει ότι θα λειτουργούν πλήρω τα ειδικευμένα δικαστήρια. Η συνεργασία του Κοσμοπεδίου με αυτά τα δικαστήρια θα είναι ζωτική σημασία για την ε, αξιοπιστία τη διεθνή του Κοσμοπεδίου και άρα για την ευρωπαϊκή του προοπτική. Ο Κοσμοπέδιο πρέπει επίση να συνεχίσει να εργάζεται με την αποστολή για το κράτο δικαίου, την ULEX, για την εφαρμογή τη εντολή τη ULEX. Αυτή είναι δέσμευση του κοσμοπεδίου με βάση τη συμφωνία. Καταλαβαίνουμε ότι η εξομάλυνση είναι προπόθεση για το κοσμοπέδιο και η πρόοδο του κοσμοπεδίου σε αυτό το τομέα είναι σημαντική για το σώμα σα η τρίτη και τελική έκθεση τη Επιτροπή για το Κοσμοπέδιο, η έκθεση πρόοδου του τελευταίου Δεκεμβρίου, σημείωσε ότι υπάρχει αξιόλογη πρόοδο, αλλά επίση τονίζει ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη πριν μπορέσει να κάνει η Επιτροπή μία πρόταση. Κάνει πολύ δουλειά το Κοσμοπέδιο για να εφαρμόσει τι ε, εναπομένουσε συστάσει και ελπίζουμε να γίνει αυτό σύντομα και τότε εφόσον έχουμε θετική έξεση, έχουμε περισσότερη πρόοδο. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για τη στήριξή σας και ε, βλέπω στην περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριάς μας είπε ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την ελληνική διερμηνία. Ελπίζω να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Αλλιώ θα πρέπει να καλέσουμε του ε, τους τεχνικούς. Ακούτε κυρία Μαριά την ελληνική διερμηνία. Μπορεί να υπήρχε κάποιο πρόβλημα προηγουμένω. Η κυρία Λούνατσεκ, η ε, συντάκτρια του ψηφίσματο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, συνάδελφε. Το Κωσυφοπαίδιο είναι η νεότερη ευρωπαϊκή χώρα. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε 8 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας ε, του Κωσυφοπεδίου σε πολύ δύσκολους καιρούς και είναι πολλοί νέοι άνθρωποι και, και φυσικά που θέλουν η χώρα τους να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρες μέλος αυτής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πρόκειται για ε, πολίτες οι οποίοι είναι υπέρ της Ευρώπης και έχουν υπάρξει πρόοδοι τα τελευταία χρόνια, όπως είπε και ε, ο Επίτροπος και ο Υπουργός. Ε, η Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση ε, ψηφίστηκε πριν από δύο εβδομάδε εδώ στην Ολομέλεια και θα τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα. Υπάρχει επίση πρόοδο ε, στο διάλογο μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβία. Δεν είναι ακόμα αρκετά φυσικά η εξέλιξη, αλλά ελπίζουμε ότι αν όλα προχωρήσουν ε, καλά, ε, θα μπορέσει το Κωσυφοπέδιο να έχει και δικό του διεθνή τηλεφωνικό κωδικό, που είναι ένα πλεονέκτημα. Αλλά δεν αρκούν όλα αυτά. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου ευθύ εξ αρχή και πρέπει να προχωρήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο, διότι η χώρα αυτή δεν αναγνωρίζεται ακόμα πλήρω από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε κράτη-μέλη ακόμα ε, αποτελούν ε, ε αναστέλουσα Δεν μπορεί να γίνει πλήρως ε, μέλος και του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα όπως για παράδειγμα την UEFA ή και το, τη Eurovision για τους θαυμαστές της ε, Eurovision. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και κυρίω ε, υπάρχει το θέμα τη απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων, όπω αναφέρθηκε. Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κλειδωμένοι στη χώρα του. Ε, ζείτε σε μία μικρή χώρα, όλοι ε, οι υπόλοιποι από τι γύρω χώρε μπορεί να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρώπη, μπορεί να επισκεφθούν την οικογένεια και τα αξιοθέατα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εσεί δεν μπορείτε παρά το γεγονό ότι οι γονεί σα και η παππούδα σα στη Ιουγκοσλαβία πάνω από 25 χρόνια πριν μπορούσαν μπορούσαν, είχαν αυτή τη δυνατότητα. Επομένως πρέπει να ε, βελτιωθεί αυτή η προσπάθεια ε, και εδώ απευθύνομαι απευθεία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου. Πρέπει να προχωρήσουν μόλις μας δώσει το πράσινο ε, φως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνω έκκληση και προς το Συμβούλιο να προχωρήσει το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων διαβατηρίων. Τώρα, για την εσωτερική κρίση στο κοσμοπέδιο. Είχαμε την, στην προηγούμενη Ολομέλεια την αντιπροσωπεία και όλες ε, οι πλευρές και η αντιπολίτευση είπαν ότι αυτή είναι η σωστή ε, ε οδός. Πρέπει να σταματήσει αυτό το μπλοκάρισμα που γίνεται στην ε, συνέλευση και να μπορέσουμε να έχουμε Ειρηνικέ ε, ε, συνεδριά χωρίς διαμάχες και πρέπει να σταματήσουν και οι διαδηλώσει στου ε, δρόμους. Και κάνουμε έκκληση και στον Πρόεδρο να βρει μια λύση για να λύσει ειρηνικά αυτή την εσωτερική κρίση της χώρας. Τώρα, όσον αφορά τι συμφωνίε διαλόγου μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου, δύο προτάσει ακόμα, κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί η συμφωνία, αλλά για να μπορέσουμε να συνδέσουμε και τους σερβικούς δήμους θα πρέπει αυτά να γίνουν με βάση και τα όσα προβλέπει το συνταγματικό δικαστήριο. Πρέπει να τηρηθεί ο νόμος ενώ η συμφωνία έχει γίνει μόνο επί της αρχής. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, τηρηθούν και τα όσα λένε οι δικαστές. Έχουμε τρεις διεθνείς δικαστές και γι' αυτό ζητώ να προχωρήσουμε και το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλές άλλες λεπτομέρειες ε, στην έκθεση, δεν μπορώ να επισέλθω βέβαια εγώ σε λεπτομέρειε το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω όλου του κοιόδη συζητητέ για την αγαστή συνεργασία και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε ε, υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, ε, ευρωπαϊκή διαδικασία τη Κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ο κύριος Αντάξουσον για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση πρόοδου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι πολύ σημαντική για το κοσυφοπαίδιο. Το Κοινοβούλιο μόλις υπερψήφισε τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Μία συμφωνία η οποία είναι όχι μόνο σημαντική για την οικονομία αλλά και για την ένταξη του κοσφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά λοιπόν αυτά τα ε, τις εξελίξεις πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Δύο παραδείγματα. Απελευθέρωση των θεωρήσεων. Πολλοί από εμάς ε, πιστεύουν ότι <clears throat> τα κριτήρια θα πληρωθούν ε, το των δυνατών. Σε τελική ανάλυση και διότι γνωρίζουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ένα σημαντικό μήνυμα προς τους κατοίκους του Κοσφοπεδίου ότι η προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει καρπούς. Δεύτερον, όσον αφορά τη σύσταση μιας ε, ένωσης ε, των ε, Σέρβων επικών, Αυτό είναι ένα από τα φλέγοντα θέματα. Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα σημαίνει περαιτέρω βήματα στον δρόμο της ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Σερβία και επιστροφή σε επικοδομητικές σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στην Πρίστινα. Κυρία Πρόεδρε, με το ψήφισμα που συζητάμε σήμερα, αυτό είναι πολύ καλά προετοιμασμένο από την κυρία Λούνατσεκ και αντικατοπτρίζει την επικρατούσα άποψη στο Κοινοβούλιο. Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την εξέλιξη, ε, το ΕΛΚ θα πει ναι στο ψήφισμα στην τελική ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την αξιότιμη κυρία Λούνατσεκ για τη δουλειά της. Αυτή η έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Κοσμοπέδιο φωτογραφίζει την τρέχουσα κατάσταση. Είναι μια μεταβατική κατάσταση και όπως ελέγχεται ήδη είναι πολύ σημαντικό το ότι υπογράφηκε η συμφωνία και θα εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Αναφέρομαι προφανώς στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, μια συμφωνία η οποία επιβεβαιώνει την ευρωπαϊκή προοπτική για το Κοσμοπέδιο κοσφοπέδιο. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι απαραίτητε συνθήκε έτσι ώστε στο Κοσμοπέδιο να υπάρξει σταθεροποίηση και αυτό να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση Λούνατσεκ δείχνει τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Πρέπει να έχουμε σταθερά βήματα προ την κατεύθυνση της ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Σερβία, να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσει, οι προσπάθειε μεταρρύθμιση εκ μέρου τη δημόσια διοίκηση είναι σημαντικέ, αλλά δυστυχώς ε, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια πολιτικά, πολιτικές εξελίξεις που δημιουργούν πολλές ανησυχίες. Υπάρχει σε επίπεδο ε, οικονομίας έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ε, μαύρη οικονομία και υψηλό ποσοστό ανεργίας. Αυτά παρεμποδίζουν την ανάπτυξη στη χώρα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με σοβαρότητα, όπως και επίσης το κράτος δικαίου, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο. Εμεί Εμείς σε όλα αυτά περιμένουμε να γίνουν βήματα προς τα εμπρός. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι εκ των όνου κάνευ να υπάρξει μια θετική προοπτική για το κοσφοπέδιο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αποκηρύξουν όλη τη βία που βιώσαμε πρόσφατα. Είναι λοιπόν απαραίτητο όλα αυτά να γίνουν για να ξεπεραστούν δυσκολίες, δυσπιστία σε αυτή τη χώρα ε, εκ μέρου πολλών που δεν έχουν αναγνωρίσει αυτό το κράτος. Εμείς όμως επιθυμούμε να το αναγνωρίσουμε ε, το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσαμπάσκης παρακαλώ. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Λούνατσεκ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ τη συνάδελφο Λούνατσεκ για την εργασία που επετέλεσε για το ψήφισμα και για τη συνολική συνεισφορά τη στην προσέγγιση του Κωσόβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω επίση ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους Κιώδη για τη συμμετοχή τους στο τελικό κείμενο του ψηφίσματος. Ε, συμφωνώ ιδιαίτερα με το κείμενο, περιέχει ε, αναφορές στα πολλά προβλήματα της χώρας και περιέχει και επικοδομητικές συστάσει. Αναφερόμαστε επίση στι εθνικέ μειονότητε και καλούμε το Κοσμοπέδιο να κάνει περαιτέρω προσπάθειε για την εγγύηση και την προστασία τη προστασία των Κοράνι και των Βουλγάρων. Αυτά τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα στι επαφέ μα με τι αντιπροσωπείε με το Κοσφοπέδιο. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να στηρίξω, η απελευθέρωση των προσκλητικών θεωρήσεων με το Κοσφοπέδιο. Εγώ και η ομάδα μου, η ΣΥΑ, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει βεβαιασμένα να απελευθερωθούν οι προξενικέ θεωρήσει πριν εκπληρώσει η χώρα όλε τι υποχρεώσει. Να μην ξεχάσουμε ότι το βαλκανικό τάγμα του ISIS αποτελείται από μαχητέ από το Κοσφοπέδιο και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοσφοπέδιο πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειές του για να αποδείξει ότι έχει υπάρξει γνήσια πρόοδο στην καταπολέμηση τη διαφθορά του οργανωμένου κλίματο κλπ. Γι' αυτό η ομάδα μας θα ζητήσει χωριστή ψηφοφορία για την απελευθέρωση των θεωρήσεων όπως σας ενημέρωσα κυρία Λούνατσοκ. Νομίζω για άλλη μια φορά ότι και η κυρία Λούνατσοκ και εγώ θεωρούμε ότι θα περάσει με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Βάουτμαντς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν χώρες που θέλουν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι που θέλουν να προσχωρήσουν περίεργος κόσμος η Ευρώπη μπορούμε να πούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λουνάτσο και την εισηγήτριά μας, γιατί εργαστήκαμε πολύ καλά και με άλλους συναδέλφους και το αποτέλεσμα λαμβάνει υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις. Στις 21, Ιανουαρίου είχαμε συζητήσεις των δύο κομμάτων που επιχείρησαν να κάνουν μια προσπάθεια προσέγγισης και γι' αυτό υποβάλαμε μια τροπολογία για το θέμα αυτό και νομίζουμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί γιατί είναι κάτι που δεν ε, περιλαμβάνεται στο ψήφισμα. Εδώ έχουν περάσει μήνες από τότε που συνάφθηκε το σύμφωνο και πριν από 15 χρόνια όταν ήμουν στα σύνορα μεταξύ Κοσμοπεδίου και Σερβίας δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τώρα έχουμε ανταλλαγές ε, φοιτητών ενώ τότε υπήρχε τόσο μεγάλη εχθρότητα. Το Κοσφοπέδιο το όντως έκανε πολύ σοβαρέ προσπάθειες και έχει και ένα όραμα, έχει προοπτικές και υπάρχουν προσπάθειες και για την ισότητα των φύλων. Όμως ε, υπάρχουν θέματα που είναι ακόμα ανοιχτά, η ελευθερία του τύπου, καταπολέμηση τη διαφθορά. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίδραση πανικού για το θέμα των προσφύγων. Και βλέπουμε ότι πολλά, πολλές δεκάδες χιλιάδες παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους θεωρούνται αγνοούμενα και πιθανώς να έχουν απαχθεί από τους διακινητές. Το κοσφοπέδιο λοιπόν πρέπει να βοηθηθεί για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ε, άθλια κατάσταση. Η Κομισιόν προτείνει φιλελευθερωποίηση των θεωρήσεων εάν εκπληρώσουμε όλα τα κριτήρια. Αυτό να το συζητήσουμε στο μέλλον. Εάν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αυτή η χώρα ε, έχει φτάσει στο αναγκαίο επίπεδο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοσομέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητάμε για την ένταξη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση του Κοσμοπεδίου. Για ένα υποτιθέμενο κράτος που δημιουργήθηκε με τις βόμβες του ΝΑΤΟ και ενθαρρύνεται από εγκληματίες που χρηματοδοτούνται από την αλβανική ε, μαφία που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους πρόσφυγες. Ας δούμε τον, εξ, ε, τον πρώην Υπουργό Τάλι που κατηγορείται για εμπόριο οργάνων από την Κάρλα Ντεπόντε και ναρκωτικών και όπλων στην ε, Χάγη θα δικαστούν αυτά τα εγκλήματα. Η αυτοανακηρυχθήσα δημοκρατία του Κοσμοπεδίου δεν ανήκει στον ΟΗΕ, δεν έχει αναγνωριστεί από την UNESCO και πάνω από 80 χώρες δεν την αναγνωρίζουν. Αλλά εξακολουθεί να ισχύει το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε στα πλαίσια αυτά να κάνει προσπάθειες ούτω ώστε να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία και όχι να αναγνωρίσει ένα υποτιθέμενο κράτος το οποίο είναι στην ουσία βήθη του αεροπλανοφόρο για τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάιο, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. εκπλήσωμε το ότι μιλάμε εδώ για την ευρωπαϊκή ένταξη του κοσμοπεδίου. Αγαπητέ συνάδελφε, μήπως θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για την ευρωπαϊκή ένταξη του συνόλου της Σερβίας. Γιατί το κοσμοπέδιο είναι ένα κομμάτι στην καρδιά της Σερβίας και η Σερβία σκόπιμα εκεί κατέστη μειονότητα. Αν δει λοιπόν κανείς τη μουσουλμανική μειονότητα στο Κοσμοπέδιο και αν θεωρήσουμε ότι δικαιούνται να ζουν σε αυτή τη χώρα, ε, τότε ε, θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες περιοχές στην Ευρώπη που δικαιούνται το ίδιο ή επιθυμούν το ίδιο. Πάντως για μας είναι σημαντικό το ότι στην περιοχή αυτή ε, κατεστράφει η σερβική ταυτότητα και αυτό είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Στον Τέτσανι, στο μοναστήρι αυτό πρόσφατα, φτυχώς προλάβαμε μια επίθεση, αλλά ξέρουμε όλο το κοσμοπέδιο ανθεί το ε, σαλαφιστικό Ισλάμ. Το ξέρουμε από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ. Κατόπιν τούτου στο, στα Βαλκάνια υπάρχουν στρατόπεδα προσιλητισμού και νεοσύλλεκτων. Αυτό δεν νομίζω ότι το θέλουμε. Ο κύριος ε, επόμενο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ κύριε Συναντινέ Βρήκε τραγέλαφο και μόνο που συζητάμε για προοπτική ένταξη περιοχή κωσυφοπεδίου μετόχια στην ευρωπαϊκή ένωση. η διεύρυνση που προωθείται με πρόσχημα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνοχή εξυπηρετεί συμφέροντα οικονομικών και γεωπολιτικών κέντρων εξουσία. α μου πει κάποιο πώ γίνεται να πραγματοποιηθεί η προσχώρηση ενό κρατηδίου όταν δεν πληρεί τα κριτήρια τη κοπεχάγη. μια περιοχή που εσκεμμένα επικίστηκε με χιλιάδε αλβανού και η οποία οραματίζεται την ένωσή τη με την αλβανία σύμφωνα με τι δηλώσει του αλβανού πρωθυπουργού ράμα και του Κοσουβάρου υπουργού εξωτερικών θάτσι πρώην ηγέτη του ουτσεκά και γνωστού εγκληματία πολέμου ενός κρατηδίου που παράγει ισλαμικό εξτρεμισμό διαφθορά εγκληματικότητα φιλοξενεί και εκπαιδεύει τζιχαντιστές και καλλιεργεί το μίσος απέναντι σε άλλους λαούς των δυτικών βαλκανίων μιας περιοχής που αποσχίστηκε βιαίως από τη σερβία και στο έδαφος της οποίας ακόμα επιχειρεί διεθνή στρατιωτική ειρηνευτική δύναμη. ήδη πέντε κράτη μέλη της ένωσης δεν έχουν αναγνωρίσει το κράτο μόρφωμα οπότε τι ακριβώς συζητάμε εδώ; ας πάψει λοιπόν η κορμοδία και ας κάνουμε το σωστό άμεση επανένωση της περιοχής κωσυφοπεδίου μετόχια με τη σερβία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση των ομιλητών εξ των πολιτικών ομάδων και τώρα περνάμε στους υπόλοιπου αγορητέ Να δώσω το λόγο στον κύριο Μακάλιστερ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη από το 2003 ισχύει το ότι και τα έξι κράτη των Βαλκανίων έχουν μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτό το υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπογραφή της Συμφωνίας Ανθρωπίσης και Σύνδεσης με το Κοσμοπέδιο, κάτι το οποίο εμείς ε, επικυρώσαμε πρόσφατα με την υπογραφή μας πριν από δύο εβδομάδες. Δυστυχώς στους δρόμους ε, της Πρίστινα και ε, άλλοι είδαμε ότι αναγκάστηκαν να φορέσουν μάσκες οξυγόνου. Αυτό επηρέασε πάρα πολύ. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, ε, τα δακρυγόνα δεν έχουν καμία θέση στο κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να υπάρχουν και να συμβαδίζουν, συμβιώνουν με τη δημοκρατία. Γι' αυτό η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν σημαντικά θέματα τη πολιτική κατεύθυνση τη χώρα. Και τέλο, να πω κάτι για τι διαπραγματεύσει με τη Σερβία. Κοιτάξτε, και οι δύο, και ο Βούτσιτ όπω και ο κ. Μούσταφα, οι δύο πρωθυπουργοί, νομίζω ότι σέβονται τις, τα ιστορικά του επιτεύγματα στι Βρυξέλλε. Οι διαπραγματεύσει ούτε ήταν ήταν ούτε είναι εύκολες. Γι' αυτό λοιπόν το Κόσοβο και η Σερβία πρέπει να εφαρμόσουν όλα αυτά που επιτεύχθηκαν. Και χαιρετίζω την ε, πρέσβη που μόλις έφτασε, όπως επίσης και την εισηγήτρια, την κυρία Λούνατσεκ. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Σάνι. Ναι. Παρακαλώ κύριε Σάνι. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε... Αγαπητοί συνάδελφοι, εξετάσαμε μια σειρά από χώρε που θέλουν να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το κοσμοπέδιο πρέπει να πούμε τα ίδια και για τις υπόλοιπες. Θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς τα καθήκοντά μας, διότι πέντε κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα να γνωρίσει το Κοσφοπέδιο σαν ανεξάρτητο κράτος. Τι νομίζετε γι' αυτό. Ο κύριος Μακάλιστερ, τα έξι κράτη των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει όλα να έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική. Έτσι αποφάσισαν το 2003 οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα έξι κράτη των Δυτικών Βαλκανίων κινούνται προ την κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια με διαφορετικέ ταχύτητε. Οπότε το θέμα τη αναγνώριση του κοσμοπεδίου είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουν κάθε κράτο μέλο κανονικά. 23 το έχουν κάνει, 5 δεν το έχουν κάνει. Εγώ είμαι από τη Γερμανία και έχουμε αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίκουλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσε για την έκθεσή της αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η υπογραφή τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση, την οποία κυρώσαμε προσφάτω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι τρόπον την αναγνώριση τη προσέγγιση του Κωσυφοπεδίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πάντα βέβαια θα εξαρτηθούν από τη συνένεση όλων των πολιτικών μερών, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Για άλλη μια φορά υπάρχουν προβλήματα στο Κοινοβούλιο, όπου κανονικά έπρεπε να είναι ο χώρο στον οποίο συζητάτε το μέλλον μια χώρα. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα χρήματα ε, προσφάτως ε, για σοβαρές ευρωπαϊκές προσδοκίες και ελπίζω τελικώς να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και το ζήτημα της ε, σύλληψης μελών της αντιπολίτευσης. το μέλλον θα είναι φυσικά η εφαρμογή όλων όσων συμφωνήθηκαν. Ε, υπάρχει υψηλό ποσοστό εγκληματικότητα, υψηλό ποσοστό ανεργία, δεν υπάρχει ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Αυτά είναι μεταξύ των θεμάτων που ακόμα ε, ταλανίζουν την κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε και τι θα γίνει με τους μετανάστες οι οποίοι πηγαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου. Ελπίζω ότι από τώρα μέχρι την επόμενη έκθεση για το κοσφοπέδιο θα έχουν επιληθεί κάποια πράγματα. Λυπάμαι που το κοσφοπέδιο δεν μπόρεσε να ε, ενταχθεί στην UNESCO. Και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα προκειμένου να ε, ε, προχωρήσουμε την άσκηση αμάλθεια ε, και κυρίως να προχωρήσουμε και θέματα που, αφορά την, που αφορούν την απασχόληση ε, και την παιδεία. Χρειαζόμαστε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και ε, το λογικό θα ήταν η νεότερη ευρωπαϊκή χώρα να έχει και ευρωπαϊκή υποστήριξη. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο κύριος Ουγιαζόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι ο Υπουργός κ. Κούντερς ε, σύντομα αλλά σαφώς εξέφρασε τι πρέπει να συμβεί στις σχέσεις μας με το κοσφοπέδιο. Πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων και επίσης να απαιτήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα προσεγγίσουν το κοσφοπέδιο στις προδιαγραφές μας. Θα προτιμούσα η έκθεση να ήταν λίγο πιο σύντομη και στοχευμένη, να αναφερθεί στα κυριότερα, για παράδειγμα, την ανάπτυξη δημοκρατικών κρατικών δομών, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καταπολέμηση της διαφθοράς και της τρομοκρατίας. Γιατί στην έκθεση αυτή υπάρχουν πολλές θέσεις οι οποίες είναι λίγο ιδεολεπτικές. Όπως και ο Σνάτο Τζαμπάσκι, θα είμαι κάπως επιφυλακτικός για την ε, ε, ταχεία απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ράντους. Ευχαριστώ πολύ. Το Κοσμοπέδιο είναι το νεότερο ευρωπαϊκό κράτος που προέκυψε από τον πόλεμο που έληξε πριν από 15 χρόνια. Το τονίζω γιατί οι χώρες που πέρασαν από πόλεμο είναι πιο δύσκολο να φτάσουν σε δημοκρατικές δομές. Είναι πιο δύσκολο να εξομαλυνθεί η κατάσταση επίσης με τους γειτονές τους. Το Κοσφοπέδιο είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντική χώρα για την εξομάλυνση των σχέσεων ε, με τη Σερβία. Και η κατάστασή του επηρεάζει τη σταθερότητα διαφόρων άλλων γειτονικών χωρών. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την υπογραφή της Συμφωνίας ε, Σταθερότητας και Σύνδεσης που θα επιταχύνει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού του κοσφοπεδίου. Και η αναγνώριση του κοσφοπεδίου από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης επίσης θα βοηθούσε. Επίσης θα βοηθούσε η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Αλλά πρώτα απ' όλα η κατάσταση στο κοινοβούλιο του κοσφοπεδίου πρέπει οπωσδήποτε να εξομαλυνθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος. Η κυρία Μπίλντε, 1,5 λεπτό. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προωθήσει κάποιες αρχές και δεν το πετυχαίνει, άρα είμαστε σύμβολα αποτυχίας, θέλουμε να ενταχθεί και ένα έδαφος που δεν έχει καμία προπόθεση για να ενταχθεί. Χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι το κοσφοπέδιο δεν είναι ανεξάρτητο κράτος που να αναγνωρίζεται από τις περισσότερες χώρες του ΟΗΕ και ιδιαίτερα πέντε χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβακία και Ρουμανία. Πολύ πρόσφατα, το 2015, 50 χώρες μέλη της Ένωσης αρνήθηκαν στο κοσμοπέδιο τη συμμετοχή ως μόνιμο μέλος. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσετε να εξηγήσετε στους Σέρβους του κοσμοπεδίου, ακόμη και αν ε, μας είπατε ότι είχατε επαφές, που υφίστανται σφαγές μεταξύ του 1999 και του 2004. 35.000 ε, σε λιγότερο από 10 χρόνια έφυγαν από τις οικίες τους. Ίσως θα πρέπει να δείξετε σε όλες τις μειονότητες, την χριστιανική μειονότητα για παράδειγμα, τη χριστιανική ορθόδοξη που διώκεται, να τους αποδείξετε πόσο καλή είναι η κατάστασή τους. Το Σαββατοκύριακο το μοναστήρι του Βιζόκη, Δεκανή, όπως ξέρετε, υπέστη νέα απόπειρα Ισλαμιστικής επίθεσης με βαρέα όπλα. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε επίσης ποια είναι τα πλεονεκτήματα να ενταχθεί στην ενωσή μας μια περιοχή όπου γίνονται κάθε είδους λαθρεμπόρια. Το 2014 ήταν στην 110η χώρα που ε, αντιμετωπίζουν καλά τη διαφθορά. Σας σέβομαι βέβαια, αλλά όταν καίγεται το σπίτι δεν ε, ε, διαμορφώνουμε τον κήπο, προσπαθούμε να σβήσουμε την πυρκαγιά. Θα ήθελα λοιπόν να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να σταματήσετε κάθε προοπτική διακόπτετη ομιλήτρια. Κυρία Μπίλντε, υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Γιάκοφτσης. Τη δέχεστε? Βεβαίως. Παρακαλώ κύριο Γιάκοβτσης. Κυρία Μπίλντε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε όπως και εγώ ότι θα ήταν καλύτερα να υπάρξει ουσιώδης πολιτική που να οδηγήσει στην ειρήνη των Βαλκανίων και όχι να υποδαβλίζουμε τις παλιές εχθρότητες και να ξεκινάμε τους παλιούς πολέμους εκ νέου. Θα ήταν καλύτερα οι δύο πρωθυπουργοί Κωσφοπεδίου και Σερβίας να ξεκινήσουν ένα διάλογο και όχι να μην μιλούν ένα τον άλλον. Γιατί έτσι θα συμβάλαμε στην ειρήνη και όχι στις διαμάχες. Και δεν θέλαμε πόλεμο. Συμφωνώ ότι οι δύο χώρες αυτές πρέπει να συνεχίσουν να έχουν επαφές. Αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα στις ίδιες μας τις χώρες σε αυτή τη συγκυρία μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο ειρηνικό κλίμα γιατί λοιπόν θέλουμε να ενταχθούν ε, στην ε, Ένωσή μας χώρες που ακόμη δεν έχουν επιτύχει κάποιο επίπεδο ειρήνευσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω το ψήφισμα για το Κωσυφοπαίδιο και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Η Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση ε, δίνει νέα προοπτική στι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κωσυφοπαιδίου. Ζητώ από το Κωσυφοπαίδιο να εκμεταλλευτεί αυτή τη συμφωνία και να προχωρήσει τι μεταρρυθμίσει που απαιτούνται για την ε, ε, ολοκλήρωση. Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται σε αρκετούς τομείς, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε και τους δημοκρατικούς θεσμούς και θέματα τα οποία σχετίζονται με το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τη διαφθορά. Διότι αυτά είναι τα θέματα τα οποία βρίσκονται στο εκεί επίκεντρο της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Ε, με εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα έχουν ε, ε, παραγωνιστεί κάπως στην έκθεση θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στο κοσυφοπαίδιο να αναπτυχθεί ώστε να μπορέσουν να νιώθουν οι Κωσοβάροι ισότιμοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με την απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων και να ε, υποστηρίξουμε και την συμμετοχή του κοσφοπεδίου σε περιφερειακές οργανώσεις. Πρέπει να αναφέρω και κάτι το οποίο αφορά την εισαγωγή της εισηγήτριας. Με όλο το σεβασμό δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπατε στην ουσία όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Λέμε στη Σερβία ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε τα πάντα ε, χωρίς ε, καμία εξαίρεση και λέμε στο Κωσυφοπαίδιο μην τηρήσετε τίποτα, μην εφαρμόσετε να περιμένετε την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Αυτά είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν μπορώ να το αποδεχθώ και θα καταψηφίσω. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Η τελευταία σας αυτή παρατήρηση αποτέλεσε πρόκληση για την κυρία Λούνατσεκ, η οποία θα ήθελε ε, μπλε κάρτα. Ε, και θα ήθελε να σας θέσει μια ερώτηση. Δέχεστε? Ναι, δέχεται ο κύριος Κούκαν. Η κυρία Λούνατσεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έντουαρτ, αγαπητέ συνάδελφε, ξέρεις πάντα ότι εκτιμώ τη συνεργασία μας, ακόμα και για το κοσυφοπαίδιο, παρά το γνωρίζω ότι η χώρα σου δεν αναγνωρίζει το κοσυφοπαίδιο, έχει επιδείξει πνεύμα συνεργασίας. Όταν όμως λες ότι στην έκθεσή μου ζητώ διαφορετικά πράγματα από αυτά που ζητάμε από τη Σερβία, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι πρέπει να κάνει η Σερβία σίγουρα πρέπει να εφαρμόσει αντίστοιχα και το κοσυφοπαίδιο. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που αφορούν το συνταγματικό δικαστήριο δικαστήριο που πρέπει να γίνουν βάσει τη συμφωνία που στις, ε, τον Αύγουστο και γι' αυτό ζητώ να υποστηρίξει και να μην καταψηφίσει την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν. Διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να σας επιπλήξω ως Πρόεδρο, αλλά παρακαλώ να διευκρινίσετε κάτι. Τώρα τι ήταν αυτό, μπλε κάρτα, ήταν ερώτημα, ήταν εισήγηση, ήταν το να μπορεί η εισηγήτρια να μιλήσει για μισό λεπτό παραπάνω στην εισήγησή τη. εντάξει το δεχτήκαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όταν θέλει να υποβάλει μια ερώτηση με μπλε κάρτα, να κάνει ερώτηση και όχι εισήγηση. Και ξέρετε, έκανε εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της. Ε, κυρία συνάδελφε, ας ε, δείχνουμε όλοι ελεγγύη προς τους συναδέλφους και ας προσπαθούμε όλοι να παραμένουμε στο χρόνο που έχει προβλεφθεί για το καθένα από εμά. Αγαπητοί συνάδελφοι, νιώθω ότι με επιπλήτεται για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγω τη συζήτηση. Κάθε φορά που κάποιος ευρωβουλευτής ε, χρησιμοποιεί μπλε κάρτα, κάνει μια ερώτηση εντός 30 δευτερολέπτων, δεν νομίζω. Βεβαίως και η μπλε κάρτα είναι για να τίθενται ερωτήσεις, αλλά περιλαμβάνει και ε, έκφραση προσωπικών απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προειδοποίηση. Η κυρία Ward, για ένα λεπτό. Χαιρετίζω τη σύσταση της συναδέλφου Λέρη και Λούνατσεκ για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, η οποία ου μόνον ενισχύει τον πολιτικό διάλογο και προσφέρει νέες μορφές συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και δυνατότητα για να ενισχύσουμε τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας και οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία με διάφορο τρόπο. Υπάρχουν πρωτοβουλίε των πολιτών που βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών στο Κωσυφοπαίδιο. Υπάρχει σεξουαλική βία από σερβικέ, στρατιωτικέ και παραστρατιωτικέ οργανώσει κατά τη διάρκεια τη σύραξη. Θα πρέπει να βρούμε επίση του μαζικού τάφου και να υπάρξει και ε, βοήθεια για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τι ζωέ του κάποιοι άνθρωποι. Πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών για να προχωρήσουν οι πολιτιστικέ ανταλλαγέ. Ε, χρειάζεται διάλογο μεταξύ των λαών και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Κωσφοπέδιου, κυρίω στην υποστήριξη των νέων ανθρώπων. Το Κωσφοπέδιο είναι η ίδια υπόσχεση για το μέλλον του. Είναι αυτοί οι οποίοι που μπορούν να κερδίσουν από το διάλογο και οι νέοι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με το ευρωπαϊκό όνομα και δεν θα πρέπει να του απογοητεύσουμε. Πρόεδρος, ε, κύριε Κιουτσούκ, επόμενος ομιλητής, ε, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Κωσυφοπαίδιο είναι η πλέον νεοκόπη ευρωπαϊκή δημοκρατία και θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ προσεκτικά τις προοπτικές της χώρας αυτής, η οποία τα τελευταία χρόνια πέτυχε πάρα πολλά και γι' αυτό οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης να θεσπίσει νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έχει επικοδομητικές ε, διαπραγματεύσεις με τη Σερβία. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχει βούληση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και για προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν η επιθυμία για αλλαγή είναι καθοριστική σημασία για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και σύνδεση που υπογράφηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία θα δώσει ότιση στην οικονομία της χώρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Κωσυφοπαίδιο πρέπει να λύσει θέματα όπως κράτος δικαίου, ελευθερία έκφρασης, αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ε, δυστυχώς δεν συμμετέχει σε όλα αυτά η κοινωνία των πολιτών. Η πρόοδος του Κωσυφοπεδίου είναι καθοριστική σημασία και για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη και έτσι λοιπόν αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από εκείνα τα κράτη τη μελη τα οποία δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του πεδίου. Πλήρη ε, ενσωμάτωση είναι η μόνη σταθερότητα για τα Βαλκάνια. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Πλένκοβιτ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Λούνετσεκ ε, για την πολύ καλή ποιοτική έκθεση. Αυτή η έκθεση θα πρέπει να αποτελεί ενθάρρυνση για την ε, περαιτέρω προσέγγιση με το κοσφοπέδιο και το χαιρετίζω αυτό όπως και τη νέα κυβέρνηση στην Κροατία. Τα λέω αυτά, ε, λέω ότι λυπάμαι που το κοσφοπέδιο δεν έγινε μέλος της UNESCO. Καλό που επιτεύχθηκε πρόοδος ε, στις σχέσεις με τη Σερβία και πρέπει να ενθαρρύνουμε την εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Η τελευταία αυτή σύνδεση και σταθεροποίηση πρέπει να βοηθήσει στο να επιληθούν ανεπίλητα προβλήματα συμπεριλαμβανομένου και του θέματος ε, των αγνοουμένων. Εγώ είμαι υπέρ της απελευθέρωσης ε, των ε, θεωρήσεων γιατί έτσι θα περιοριστεί η παράτυπη μετανάστευση. Επίσης χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις συζητήσεις σχετικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι οι συζητήσεις ε, θα είναι πολύ καλή ποιότητα στο κοσφοπέδιο και θα πληρούν και τους ε, δημοκρατικούς, ε, τα κριτήρια των δημοκρατικών θεσμών. Επόμενη μιλήτρια για ένα λεπτό. Η κυρία... Ο κύριος, με ο κύριος Βιώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα τη συνάδελφο κυρία Λούνατσα και την πολύ καλή δουλειά που έκανε η κυρία Λούνετσεκ επεξεργάστηκε το θέμα που συζητάμε σήμερα. Πρόκειται για τη θέση εφαρμογή τη τελευταία συμφωνία. Πολύ σημαντικό το βήμα αυτό για το κοσυφοπαίδιο. Ε, σημαντικό για τι μεταρρυθμίσει και για την ενίσχυση τη συνεργασία σε πάρα πολλού τομεί. Βέβαια, αυτό που ζητάνε οι κάτοικοι του Κοσοπεδίου είναι ένα πράγμα. Απαιτούν, ζητούν την απελευθέρωση των θεωρήσεων, κυρίω προ τι χώρε Σέγγεν, προ εμά. Ε, είναι σημαντικό το ότι μιλάμε τώρα γι' αυτό. Ε, το Κωσυφοπαίδιο είναι η μόνη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που δεν έχει ακόμα απελευθέρωση θεωρήσεων και είναι ε, αυτό απογοητευτικό. Όταν είχαν Ιουγκοσλαβικό διαβατήριο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Εντάξει το Κωσυφοπαίδιο πρέπει ακόμα να κάνει πολλά προς το κράτος δικαίου, προς την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό είναι η δουλειά όμως του Κοινοβουλίου. Να επαγρυπνά έτσι ώστε να χορηγηθούν δικαιώματα στους κατοίκου του Κωσυφοπαιδίου και το Κωσυφοπαίδιο να προβεί που οφείλει να εφαρμόσει. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, ο κύριος Τόκες, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για το νέο κράτος του Κοσφοπεδίου έχει μεγάλη σημασία το ότι κατάφερε να υπογράψει αυτή την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης τον περασμένο Οκτώβριο. Όμως η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έχει σημειωθεί από αυτό το κράτος της πρώην Ιουκοσλαβίας. Άρα θα ήταν λογικό να περιμένουμε παρόλα αυτά ότι και τα τελευταία πέντε κράτη-μέλη θα αναγνωρίσουν το κοσμοπέδιο και η Σερβία θα αποκτήσει ομαλές σχέσεις μαζί του. Θα ήταν επίσης λογικό να περιμένουμε το αλβανικό κράτος, αυτό το νέο κράτος, να κάνει όλες τις αναγκαίες ε, προσπάθειες για να καταπολεμήσει τη βία και τη διαφθορά. Πρώτα απ' όλα η νέα κυβέρνηση πρέπει να χορηγήσει τα δικαιώματα που είχε δικαίως απαιτήσει από την ε, προηγούμενη σερβική πλειοψηφία η ίδια να τα χορηγήσει αυτά σερβική μειονότητα. Στην πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Κοσφοπέδιο και η Σερβία αλληλοεξαρτώνται. Είναι δική τους επιλογή αν θέλουν να αλληλοϊποστηριχθούν. Μόνο έτσι όμως θα ενταχθούν. Γιατί αλλιώ απλώ θα μπλοκάρουν ένα τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μαμίκιν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, από τότε που το 2008 διακήρυξε μονομερό την ανεξαρτησία του, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν αμέσω ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξη του Κοσμοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει ότι στην ουσία είναι οι κύριοι διαπραγματευτέ μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Αυτό σημαίνει ότι αν το κοσμοπέδιο θέλει να γίνει μέλος της οικογένειας εθνών μας, πρέπει να σεβαστεί τις αξίες μας. Δημοκρατία, ελευθερία λόγου, καλή διακυβέρνηση, όλα αυτά πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστά. Αυτό δεν είναι προαιρετικό, είναι υποχρεωτικό. Δεύτερον, το κοσμοπέδιο και η Σερβία πρέπει να φτάσουν σε έναν αμοιβαία αποδεκτό συμβασμό, ούτως ώστε να υπάρξει μακροπρόθεσμα ειρήνη και συνεργασία. Η στάση των Σέρβων έναντι του κοσμοπεδίου είναι ότι είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι γιατί έχασαν την ιστορική τους κοιτίδα. Η αλληλοκατανόηση πρέπει να λύσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει προοπτική ένταξη του κοσυφοπεδίου αν δεν το αναγνωρίσουν όλα μα τα κράτη-μέλη ω ανεξάρτητο. Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ισπανία, πέντε από τα 28 κράτη-μέλη δεν το έχουν ακόμη κάνουν. Ο καθένα για του λόγου του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πέτερλε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κοσφοπέδιο με αυτή τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λούνατσεκ για άλλη μια θαυμάσια έκθεση που εξεπώνησε. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει το κοσφοπέδιο να προχωρήσει ακόμη περισσότερο γιατί δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση στην ειρηνική συνύπαρξη με βάση βέβαια την ε, αναγνώριση των αρχών της ταυτότητας και όλων των δικαιωμάτων όλων των ε, τμήματων του πληθυσμού. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προσπάθειες που έχει κάνει η κυρία Μογκερίνη προς αυτή την κατεύθυνση. Και πρέπει να δούμε και πώς θα λύσουμε το θέμα της ε, φιλελευθερωπήσης των ε, θεωρήσεων στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άσης για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν θα πρέπει να ε, ξεχνάμε ότι οι αρχές του Κωσυφοπεδίου είναι και αυτές σε διαπραγμάτευση υπέρ της ειρήνης και ενδιαφέρονται για τις σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Στη διαδικασία ε, προσχώρησης της ε, ε, το Κοσμοπέδιο αποδεικνύει ότι παραμένει ζωντανό το ευρωπαϊκό όραμα παρά την κρίση. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Μογκερίνη, η οποία προσπάθησε να εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας και να την ευχαριστήσω γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση μεταξύ των Σέρβων και των Κωσοβάρων. Η πορεία ε, βέβαια ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μια προοπτική στο κοσφοπέδιο, διότι ε, αλλιώς ε, θα τους απογοητεύσουμε. Ε, πρέπει να προωθήσουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση του λαού και να μπορέσει να προσεγγίσει το κοσφοπέδιο την Ευρώπη. Με αυτό ολοκληρώνεται ο κατάλογος των αγορητών. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ, αλλά θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα πέντε λεπτά. Η κυρία Σουίτσα, καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την ιδιαίτερα ποιοτική έκθεσή τη. Αλλά να ευχαριστήσω και την κυρία Μογερίνη και τον κύριο Χάν, οι οποίοι έχουν εργαστεί σκληρά ώστε να μπορέσουμε και εμείς ε, να ε, αξιολογήσουμε την έκθεση προόδου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Η σταθεροποίηση του κοσυφοπεδίου είναι καλή για τη σταθεροποίηση όλη τη περιοχή των Βαλκανίων. Το πιο σημαντικό στοιχείο βέβαια είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία. Έχουν γίνει πάρα πολλά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει ακόμα να γίνουν αρκετά περισσότερα και να ζητήσουμε περισσότερα. Πρέπει η Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και επίση πρέπει να βελτιωθούν και οι σχέσει μεταξύ τη ε, κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση. Ε, είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ενταχθεί στην UNESCO το κοσφοπέδιο και ε, είναι κρίμα που ε, χρησιμοποιείται η κατάσταση ως ένα μέσο εκβιασμού. Πιστεύω ότι οι πέντε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο θα πρέπει να το κάνουν τώρα. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, το Κόσοβο αποτελεί άλλο ένα θλιβερό τερατούργημα στρατιωτικών επεμβάσεων στις οποίες συνέδραμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνουμε ότι το ψευδοκράτος του κωσόβου έχει μονομερώς κηρύξει την ανεξαρτησία του που είναι αντίθετη με το ψήφισμα 1244 του συμβουλίου ασφαλείας του οηε το οποίο προβλέπει αυτονομία του κωσόβου εντός της σερβικής επικράτειας. σημειώνουμε επίσης ότι σε σχετική έκθεση του συμβουλίου της ευρώπης ο νυν υπουργός εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός του ψευδοκράτους χασίμ θάτσι κατηγορείται για σύσταση δικτύου παράνομης εμπορίας ανθρώπινων οργάνων επισημαίνουμε τους συστηματικούς διωγμούς και απειλές που βιώνουν οι χριστιανοί του κωσόβου στην πλειοψηφία του σέρβοι. σημειώνουμε ότι το κόσοβο βρίσκεται στη λίστα των δέκα κρατών με τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που εμπλέκονται άμεσα στην ισλαμική τρομοκρατία του νταές σημειώνουμε επίσης ότι το εθνικιστικό κίνημα που διεκδικεί ένωση με την αλβανία λαμβάνει το 14% των ψήφων. στα στοιχεία λοιπόν αυτά δείχνουν ότι είναι απαγορευτικά για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πορεία ενός κράτους παρία που άλλωστε δεν την χάνει αναγνώρισης από το σύνολο των κρατών της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. χωρίς ε, τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων δεν μπορούμε να φανταστούμε ε, μια ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοσμοπέδιο πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά φυσικά ε, απομένουν πολλά ακόμα. Θα ήταν χρήσιμο τα υπόλοιπα πέντε κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν και αυτά το Κοσμοπέδιο. η απόσχεση του Κοσμοπεδίου από τη Σερβία δεν έγινε ομαλά. Αντίθετα, Αυξήθηκε, οι ε, περιφερειακές αυτονομίες μειώνουν τις εντάσεις μεταξύ εθνικών μειονοτήτων και οδηγούν προς την ειρήνη. Το κοσφοπέδιο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πόσο κακή τροπή μπορούν να πάρουν τα πράγματα εάν δεν υπάρχει ε, προσοχή. Ε, αυτό είναι ένα επικίνδυνο λοιπόν προηγούμενο απόσχεσης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω, να ζητήσω κάτι. Η προηγούμενη πρόεδρος μου έδωσε μπλε κάρτα και θα ήθελα να παρακαλέσω αν μπορεί ο κ. Σελίμοβιτς να μιλήσει εκ μέρους μου, να με αντικαταστήσει μάλλον, ομιλώντας εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης ε, και το συνάδελφο. Η προσέγγιση του κοσμοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το θετικό, έτσι Έχουμε ένα τέλος στη σύγκρουση στο κοσυφοπαίδιο και βεβαίως ε, θα υπάρξει βελτίωση μόνο εφόσον εφαρμοστούν ταχύτατα οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το θέμα της σερβικής μειονότητας πρέπει να επιληθεί, όπως επίσης και η αναγνώριση του κοσυφοπαιδίου και η ομαλοποίηση των σχέσεων με τη χώρα αυτή. Αυτά είναι προϋπόθεση για την ε, προσέγγιση με τη Σερβία. Ε, και αυτά είναι και προαπαιτούμενα για το κοσυφοπαίδιο με την έννοια ότι πρέπει να λύσει το θέμα της σερβικής μειονότητας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι προσπάθειες μιας νόμιμης κυβέρνησης να αφαλκιδεύονται από την αντιπολίτευση. Στην περίπτωση αυτή ε, θα πρέπει και η αντιπολίτευση να τοποθετηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο κύριος Στόλτας. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την ε, θαυμάσια έκθεση της στο Κωσοφοπέδιο. Είναι από τις νεότερες δημοκρατίες και είναι ένα κράτος με νεότατο πληθυσμό. Από εμά λοιπόν εξαρτάται εάν η χώρα αυτή θα μπορέσει να γίνει μια κανονική δημοκρατική χώρα με αναπτυγμένους ε, μηχανισμούς για να αποφύγουμε μαζική μετανάστευση και για να αποκτήσει μια προοπτική. Πρέπει φυσικά να γίνουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να εξηγιανθούν τα δημοσιονομικά και να αναπτυχθούν καλές σχέσεις γειτονίας με τη Σερβία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει το κοσφοπέδιο να γίνει πραγματικά ανεξάρτητο και να γίνει μέλος πολλών σημαντικών διεθνών οργανισμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω κάνει διάφορες ερωτήσεις προς την Κομισιόν για εδάφη που θέλουν αυτοδιάθεση και ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τα διεθνή και τα διεθνώς αναγνωσμένα σύνορα. Τώρα εδώ δεν τα αναγνωρίζει όμως. Δεν είναι υποκρισία αυτό παραβιάζουμε τους δικούς μας κανόνες. Ε, τα μέσα αιτιολογούν το σκοπό. Το κοσμοπέδιο δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος από τα Ηνωμένα Έθνη, όμως έχουμε πολύ αναπτυγμένες σχέσεις και το αναγνωρίζουμε ως ενδεχόμενη υποψήφια χώρα. Παρά το ότι δεν υπάρχει βιώσιμη πολιτική λύση μεταξύ της Σερβίας και του Κοσφοπέδιου. Και αυτή η ιδιαίτερα παρεμβατική ε, διπλωματία μας στην ουσία αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή θα τα κάνει όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την νεοαπικιακή της ε, στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόλτσακ. Δεν είναι παρόν. Ο κύριος Ομπεμάερ, τελευταίος. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω να λέμε τα πράγματα με το όνομά τη. 200 ε, ε, τζιχαντιστέ, ένα εκατομμύριο. είναι η αναλογία ε, στο Κωσυφοπαίδιο. Και αυτό ξεπερνάει και το Βέλγιο και ξεπερνάει και το ποσοστό στη Λιβύη. Δηλαδή στη χώρα αυτή έχουμε τζαμιά από σκληροπυρηνικού Ισλαμιστέ. Το Κωσυφοπαίδιο δεν έχει καμία σχέση με το λαϊκιστικό Ισλάμ όπω το γνωρίζαμε. Γι' αυτό λοιπόν μια ελβετική εφημερίδα προβλέπει ρεαλιστικά ότι το Κοσμοπέδιο θα είναι το πρώτο Ισλαμικό κράτο, θα μπορούσε να είναι το πρώτο Ισλαμικό κράτος Ευρωπαϊκή Ένωση. Συν τη άλλη το Κοσμοπέδιο είναι ο κόμβος τη διεθνού εγκληματικότητα. Ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ε, να πούμε για ένωση με αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχουν ούτε κοινωνικοί ούτε πολιτικοί λόγοι. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σεβαστή η βούληση των ε, Ευρωπαίων πολιτών που δεν θέλουν Ισλαμικό κράτο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσωπικά φοβάμαι ότι με το Κωσοπέδιο θα έχουμε, θα βάλουμε μόνοι μας σε λειτουργία την επόμενη ευρωπαϊκή ορολογιακή βόμβα. Τελείωσε η διαδικασία Catch the Eye, λέει η πρόεδρος και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Χάν για να εξάγει τα συμπεράσματα του εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ στο Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι όσον αφορά στην ε, ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκονίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρειαζόμαστε αυτό ε, και η οικονομική ανάπτυξη τη περιοχή αυτή ε, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα σήμερα ε, κάποιο εκνευρισμό εκ μέρους κάποιων συναντέλφων και θεωρώ ότι αυτό θα διαλυθεί μόνο εάν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε και για στρατηγικούς πολιτικούς λόγους το να υπάρχει ένα κενό, μια μαύρη κοιλίδα στα Δυτικά Βαλκάνια όπου δεν θα ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, δεν θα υφίστανται οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες και ε, ίσως αυτό να έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες. Άρα δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη αυτών των κρατών. Ε, σαφές ότι ε, δεν μπορούμε να πάμε εκεί όπου θέλουμε ή τίποτε το θέλουμε. Νομίζω όμως αυτή τη διαδικασία έχουμε μια διαδικασία που ξεκινάει. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα αυτή στην οικονομική της ε, ανάπτυξη, ε, στα νομοθετικά της προγράμματα, να τη φέρουμε κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Κοσμοπέδιο αυτή η τελευταία συμφωνία σύνδεσης και σταθεροποίησης είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο, το πλέον ενδεδειγμένο εργαλείο και αυτό που έχει τώρα σημασία είναι η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Απευθύνομαι λοιπόν σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του κοσμοπεδίου να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Έχουμε πλήρη κατανόηση για πολιτικές αντιπαρατέσεις. Εξάλλου το έχουμε συνηθίσει όλοι μας αυτό εδώ όλοι μας αυτό όσοι βρισκόμαστε εδώ. Υπάρχουν όμως κοινοί εθνικοί στόχοι και δεν νομίζω ότι πρέπει να τους αφαιρέσουμε την πολιτική προοπτική γιατί αυτή θα ενώσει την πλειοψηφία. Ως εκ τούτου εγώ απευθύνομαι στους αρμόδιους στο Κοσμοπέδιο, κάνω έκκληση να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι και μέσα από τη συζήτηση να θέσουν τα θεμέλια για την πολιτική εξέλιξη της χώρας να αποκηρύξουν οποιαδήποτε μορφή βίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαρασάλευτα θα συνεχίσει να προσπαθεί να φέρει κοντά το κοσμοπέδιο στην ευρωπαϊκή προοπτική. Απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ήδη αναφέρθηκε αυτό. Η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Κυρίε και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι το κοσυφοπέδιο πάνω από ένα τρίτο των εσόδων του το εισπράττει από σε μια Ευρώπη χωρίς δασμούς. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ήδη τώρα να ξεκινήσουν σιγά σιγά να τα αλλάζουν τα πράγματα έτσι ώστε να ε, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Υπάρχει και το θέμα της υψηλής ε, ανεργίας, ε, μια τάση που διαφαίνεται σε αυτή την περιοχή. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν τα μέτρα που προανέφερα. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε έτσι ώστε στην περιοχή αυτή να επικρατήσουν ειρήνη, σταθερότητα, προοπτικές για τους ανθρώπους έτσι ώστε να μείνουν και αυτοί εκεί, σε αυτή την περιοχή και να μην είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος υπουργό έχει το λόγο για να ε, ολοκληρώσει εκ μέρους του Συμβουλίου. Uh, Ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ευγενή μου ε, την ευγνωμοσύνη μου συγγνώμη, στην ε, εισηγήτρια την κυρία Λούνατσεκ που εκπώνησε την έκθεση αυτή για το κοσφοπέδιο. Ξέρετε ότι το κοσφοπέδιο έχει ένα παρελθόν ε, πολλή βία, το ανεφέρετε αρκετοί από εσά και νομίζω ότι ορθά μιλήσατε. Αν δείτε την κατάσταση από το 1999 έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος και πρέπει να το ενισχύσουμε. Έχει σκαμπανεβάσματα βέβαια η διαδικασία, αλλά ε, σας δηλώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συνδράμει το κοσφοπέδιο και με παρουσία επιτόπου και φυσικά η βασική ευθύνη για την πρόοδο με το κοσφοπέδιο, με τους ηγέτες της, με τα ε, θεσμικά όργανα τη και με την κοινωνία των πολιτών είναι προτεραιότητές μας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει οι επικεφαλείς ε, να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων για το καλό των πολιτών του Κωσφοπεδίου και επίση ε, ε, θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσει όχι για να ευχαριστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι προ το συμφέρον τη ίδια τη χώρα. Όσον αφορά την πολιτική κρίση σίγουρα παρακολουθούμε με ανησυχία την ε, κατάσταση όπω και αρκετοί από εσά. Έχουμε διευκρινίσει ότι η βία δεν είναι αποδεκτή για πολιτικού σκοπού και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα μέσω κοινή προσπάθεια και πολιτικού διαλόγου. Η συγκήτρια νομίζω αναφέρθηκε και στο Συνταγματικό Δικαστήριο του Κοσφοπεδίου. Όπως γνωρίζουμε αποφάνθηκε ότι η Ένωση των Σερβικών Δήμων θα πρέπει να συσταθεί όπως προβλέπεται από την πρώτη συμφωνία βάσει και του Συντάγματος και φυσικά θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε ε, με τη σύνταξη του, ε, του καταστατικού της Ένωσης για να προχωρήσει αυτός ο διάλογος. Αναφερθήκατε επίσης και στις ευρωπαϊκές προσδοκίες ε, των πολιτών του Κοσμοπεδίου. Άκουσα βέβαια και το τι δήλωσαν και κάποιοι από ε, την ε, συγκεκριμένη πλευρά που αναφέρθηκαν σε αντιισλαμικά φρονήματα και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει τέτοιο λεξιλόγιο. Θα πρέπει να περιοριστείτε σε επιχειρήματα τα οποία σχετίζονται με την ίδια την υπόθεση και να μην οδηγείτε, οδηγείστε σε σχόλια τα οποία οδηγούν σε διακρίσεις. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και μια ευρωπαϊκή προοπτική για το κοσμοπέδιο, αλλά όπως είπε και η κυρία Λούνατσεκ υπάρχει πρόοδος αλλά δεν αρκεί. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολλά προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση και φυσικά αυτό θα δώσει ελπίδα στους νέους ανθρώπους. Ε, χρειαζόμαστε απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων ε, και θα μπορούν έτσι οι νέοι να ταξιδέψουν, αλλά χρειαζόμαστε και την καταπολέμηση της διαφοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, ε, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις εκ των νόνου κάνευ για να προχωρήσει η διαδικασία θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε το Κοσμοπέδιο και με χρηματοδοτική στήριξη και μέσω εμπειρογνωμοσύνης, μέσω της EULEX και φυσικά εάν ε, έχει αποτελέσματα το Κοσμοπέδιο θα μπορέσουμε και εμείς ε, να ε, προχωρήσουμε με τις δεσμεύσεις μας. Αυτό ελπίζω ότι θα σημαίνει ότι θα μπορούν οι κάτοικοι του κοσφοπεδίου να ταξιδεύουν ελεύθερα όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Κάτι τελευταίο, να σταθώ στη σημασία της θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας και σύνδεσης μετά την κύρωση από πλευρά σα. θα πρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει τα συμπεράσματά του ε, υπάρχει τέτοιο προγραμματισμός και από εκεί και πέρα θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο μήνα μετά την κοινοποίηση και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε από 1η Απριλίου ή από 1η Μαΐου να ε, ξεκινήσουμε με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έτσι λίγη συζήτηση για το θέμα αυτό. Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσμα.